Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίσω την έναρξη των εργασιών της δεύτερης αυτής συνεδρίασης της κοινή Επιτροπής για το σχέδιο προπολογισμού για την Ευρωζώνη. Η Υπερβάνος Μπερές, που είναι συνεισηγήτρια, μαζί με τον Ράιμερ Μπέγκε, θα έλθει εντός ολίγων λεπτών Παρ' όλα αυτά προτείνω να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Οι δύο εισηγητές έχουν υποβάλει ένα δεύτερο έγγραφο εργασίας. Το δε σχέδιο έκθεσής τους ε, θα είναι έτοιμο μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Θα ακούσουμε λοιπόν τους δύο εισηγητές και στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο οι σκιώδεις από τις επιτροπές Έκον και Ο Ράιμερ Μπέγκε. Eh bien, la parole est à Ja, vielen Dank, äh, meine Herren Vorsitzenden, äh, liebe Kollegen. Ευχαριστώ αγαπητοί πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά ε, προετοιμάσαμε το έγγραφο εργασίας και υπό το φως των παρουσιάσεων που ακούσαμε και με βάση τα όσα είχαν ε, εντωμεταξύ πει οι ομάδες. Θα ήθελα να πω επί της αρχής ότι αν είδε κανείς μια συνέντευξη του Μάριο Μότι αυτή της εβδομάδας που σας διαβάζω φοβάται ο Μόντι ότι η εθνική διαφθορά, οι μηχανισμοί των Βρυξελών και ο συνδυασμός τους μπορεί να οδηγήσουν σε κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει ξαναμιλήσει νομίζω τόσο ανοιχτά ο Μάριο Μόντ και έχει δίκιο εδώ πέρα γιατί το θέμα του πόσων μας ενώνουν σε αξίες και αρχές ε, βρίσκεται στις ε, συμβάσεις που έχουν υπογράψει τις τηρούμε ή είμαστε σε κάποια τμήματα του δυτικού κόσμου σε μια πορεία εθνικισμού και λαϊκισμού και τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Πρέπει να μας ανησυχήσει αυτό. Και αυτό σχετίζεται με το θέμα το οποίο έχουμε να συζητήσουμε σήμερα για τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές δυνατότητες. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον και ένα τέτοιο κλίμα. Είναι λογικό να πούμε ακριβώς επειδή εκτιλήσεται έτσι η συγκυρία και επειδή πάρα πολλοί πολίτες από ανησυχία για την προσωπική τους κατάσταση εξισώνουν την Ευρώπη με κάποιες ε, πιέσεις που υφίστανται λόγω της παγκοσμιοποίησης και θεωρούν την Ευρώπη κομμάτι της παγκοσμιοποίησης και όχι κομμάτι της λύσης. Εμείς θα κάνουμε λοιπόν. Θα καθόμαστε να κοιτάμε ή θα αντιδράσουμε και θα προτείνουμε ενεργητικές ε, λύσεις ε, παρόλη την αντίδραση για να υπάρξει μια σταθεροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών. Αυτό το βασικό ερώτημα πρέπει να απαντήσουμε όταν ρωτάμε ποια στρατηγική θέμε να ακολουθήσουμε. Οπωσδήποτε είναι θεμητό να πούμε πως χρειαζόμαστε πολλά μικρά ε, βήματα που τελικά και αυτά οδηγούν στον στόχο μας. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι εάν έχουμε χρόνο πια. Έχουμε πολλές κρίσεις τις οποίες εγώ δεν έχω ξαναδεί στην πολιτική μου ζωή να συμπίπτουν χρονικά και κάνουν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά αν δεν κάνουμε τίποτα, τότε σε δύο-τρία χρόνια θα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση είτε διάλυσης ε, είτε ανάγκης ε, επανίδρυσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήθελα λοιπόν να τα πω αυτά γνωρίζοντας πως ε, κάποια από τα πράγματα τα οποία θα πούμε δεν θα δημιουργήσουν και άκρα τη χαρά στα κρατημέρια, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να τα πούμε. Έχουμε λοιπόν ένα έγγραφο εργασίας το οποίο αναδεικνύει μια σειρά ερωτήσεων και θα ήθελα να ζητήσω να δω και να ρωτήσω βέβαια στους υπεύθυνους των ομάδων γιατί χρειάζονται κάποια πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε για δημοσιονομική δυνατότητα. Γιατί χρειάζεται δημοσιονομική δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε ποια μέσα έχουμε αυτή τη στιγμή σήμερα με τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία συνοχής, ε, το ΕΦΣΥ, τη γεωργία. Φτάνουν αυτά ή μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και δουλειές. και να μπορέσουν μετά και οι χώρες να ακολουθήσουν και τις συστάσεις ανά χώρα. Νομίζω λοιπόν πως ένα βασικό ε, ερώτημα για να υπάρξει αποδοχή των περαιτέρω βημάτων είναι αυτό. Το θέμα των λειτουργιών μιας δημοσιονομικής ικανότητας. Για να το ξεκαθαρίσω. Εγώ και νομίζω και οι περιβάλλοντες εδώ πέρα θα συμφωνήσει πως ο στόχος είναι η εσωτερική αγορά και το νόμισμα είναι το ευρώ. Τα υπόλοιπα είναι εξαιρέσεις και οι χώρες οι οποίες ε, αυτή τη στιγμή έχουν μία εξαίρεση κάποια στιγμή θα μπουν στο ευρώ. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να δούμε τα όσα αναφέρονται στι συμβάσει που έχουν υπογράψει και τα όσα μα ενώνουν και δεν μα διαχωρίζουν. Έχουμε λοιπόν αυτά τα υφιστάμενα μέσα και με τα δικαιώματα συναπόφαση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δημιουργία λοιπόν μια δυνατότητα προπολογισμού για την Ευρωζώνη, συμπληρωματική και όπου και αν εδράζεται αυτή, έχει έναν κίνδυνο και τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή κύριε Πρόεδρε. Έχουμε το outsourcing των trust funds. Δηλαδή, η δουλειά του Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή ανατίθεται σε άλλους εξωτερικούς και υπάρχουν ε, δομές οι οποίες αναπτύσσονται και ακριβώς αυτός είναι και ο κίνδυνος εδώ πέρα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό λοιπόν γιατί το θέμα του πόσες επιδοτήσεις λαμβάνει κάποιος για επενδύσεις ή δεδομένων των επιτοκίων σήμερα το θέμα δεν είναι μόνο να δώσουν περισσότερο κίνητρα με δημόσιο χρήμα αλλά πρώτα απ' όλα όπως το είχε πει και ο Λούτβι Χέρχαρτ τότε στην Γερμανία αυτός ο οποίος ε, έστησε την μεταπολεμική γερμανική οικονομία είχε πει ότι πάνω από 60% της οικονομίας είναι η εμπιστοσύνη η πίστη. Έχοντας πει αυτά λοιπόν θα ήθελα να πω το εξής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε άμεσα από τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται αλλαγή των συνθήκων. Παραδείγματο χάρη υπάρχει αυτό το οποίο πρότεινε ο καθηγητής ε, ο Άξονεν για ένα σύστημα ασφάλειας, ασφάλειας των καταθέσεων το οποίο θα είναι και δίκαιο για να στείλουμε ένα ε, μήνυμα αλλά ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει να πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσω με τις αναγκαίε προσαρμογές και τελικά γιατί δεν μιλάμε όταν βλέπουμε τον ESM και βλέπουμε πως ε, εντωμεταξύ η κατάσταση του δικαίου βρίσκεται σε μια ελεύθερη πτώση. Π.χ. έχουμε το άρθρο 143, το οποίο χρησιμοποιούν χώρες εκτός της Ευρωζώνης με 3 και 4 δισεκατομμύρια μετά έχουμε το άρθρο 122 παράγραφος 2, το οποίο προσπαθήσαμε, δηλαδή το κοινοβούλιο σε μια μεγάλη νύχτα βρέθηκε εκτός και αποφασίστηκε το ESM να ε, εκταμπιεύσει 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο. Ήταν μια επίθεση στα δικαιώματα του Κοινοβουλίου και το διορθώσαμε και το βάλαμε στη διαδικασία του υπερπολογισμού. Και τώρα έχουμε το ESM που είναι διακυβερνητικός μηχανισμός γιατί προφανώς δεν γινόταν αλλιώς. Βλέπουμε την εξέλιξη όμως. Η τάση που υπάρχει σε όλα αυτά τα πράγματα είναι αρνητική για την κοινοτική μέθοδο. Δεν σημαίνει πως η κοινοτική μέθοδος θα κάνει όλα καλύτερα, γιατί και εκεί πέρα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνοηθούν κάποτε, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε πως υπάρχει ένα νομισματικό ταμείο και στην Ασία όπου οι χώρες βάζουν κάποια λεφτά στην άκρη για να βοηθηθούν σε καιρούς κρίσης. Και εδώ πέρα δεν κατηγορώ το ΔΕΛΤΑΝΤΑΦ. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να ενσωματώσουμε κάπου τις σκέψεις 2010, του 2010-2011, δηλαδή το ESM να μεταβληθεί σε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο, κάτι το οποίο όμως σημαίνει ότι θα υπάρχουν συνταγματικές αλλαγές για να λειτουργεί με τρόπο αξιόπιστο. Δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε ένα θέμα Υπουργείου Οικονομικών, ένα θέμα οικονομικής διακυβέρνησης και λοιπόν αλλαγών. Αν είναι να είμαστε δηλαδή αξιόπιστοι. Και βεβαίω τίθεται και το θέμα της ε, ευθύνη που θα έχει ένα τέτοιο Υπουργείο Οικονομικών για την Ευρωζώνη και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει και προβλεπόμενη διαδικασία μιας κρατικής χρεοκοπίας ως τελευταία επιλογή εάν κάποιες χώρες δεν τηρούν τους κανόνες. Μόνο ως πακέτο μπορούν να γίνουν αυτά και βεβαίως να συζητήσουμε μετά τι χρειαζόμαστε ως δημοσιονομικές δυνατότητες, ως δημοσιονομικές δυνατότητες για να σταματήσουμε ή να αντιμετωπίσουμε τα σοκ και εδώ πέρα βλέπω μια θετική εξέλιξη σταδιακά στο Συμβούλιο, αν διαβάσατε τη συνέντευξη του Φίλιπ Μάιστατ, που είχε πει πως υπάρχει στήριξη και κλεισμένων των θυρών για τους όρους, ε, για την αίρεσιμότητα των προγραμμάτων κάποιων χωρών που είναι σε δυσκολίες. Για να δουν μετά υπό ποια μορφή θα μπορέσουμε να πάμε σε μια τέτοια δημοσιονομική δυνατότητα, αν θέλετε πείτε το ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο γιατί ε, βεβαίω θα πρέπει να δούμε και την τάξη των ε, μεγεθών που είναι διατεθειμένα να διαθέσουν το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Αυτά κύριε Πρόεδρε θα ακούσετε βέβαια και την συνεισηγήτρια μου. Ευχαριστώ τον Ράιμερ Μπέγκε. υπέρ μας Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη για την ε, καθυστέρηση. Αλλά είχα κάποια προβλήματα στο Παρίσι. Έχουμε ξεκινήσει, από τότε επαναλάβαμε αυτήν την βαριά ευθύνη το έργο μας για να ξεκινήσει ενδεχομένω μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έναν προπολογισμό της Ευρωζώνης από Ακούσατε, είχαμε κάποιες διαβουλεύσεις, οργανώθηκε και μία ακρόαση από τους δύο προέδρους ε, των ε, συναρμοδίων επιτροπών και ακούσαμε απογοητευτικά ε, και από το Δέλτα Νιτάφ, από τον διοικητή της Τράπεζας των Κάτω Χωρών και το διοικητή ε, της Παγκόσμιας Τράπεζας. Διότι ο Ράιμερ ε, Μπέγκε, και συμφωνώ μαζί του, παρότι δεν έχουμε ε, ψευδεστήσεις, γνωρίζουμε ότι ένας ειδικός προπολογισμό για την Ευρωζώνη μπορεί να ήταν κάτι λανθάνων μετά την ΟΝΕ αλλά και μετά το blueprint του 12 είναι ξεκάθαρο και οι αναλύσεις που έχουν γίνει έκτοτε επιβεβαιώνουν ότι λείπει ένας πυλώνας από την ΟΝΕ, ο συγκεκριμένος πυλώνας. Το πλαίσιο σήμερα έχει ως εξής. Υπάρχει ακαδημαϊκός προβληματισμός, σημαντικός μέχρι τώρα. Δεν έχουμε βέβαια εξαντλήσει το θέμα. και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε τι συνιστά οικονομικό, οικονομική συλλογιστική και τι εμπίπτει στο πολιτικό επίπεδο. Και πρέπει να βρούμε το πού τέμνονται και ποιος είναι ο κοινός χώρος μεταξύ των δύο. Αυτή η έκθεση δεν είναι μετέωρη. Έχει προηγηθεί, όπως είπα, και προβληματισμός γενικότερος. Είχαμε και την ευθύνη για την έκθεση περί Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης. Οπότε, στο πλαίσιο αυτό, δώσαμε έμφαση στις ανεπάρκειες της ΟΝΕ και ιδίως στο γεγονός ότι δεν λαμβάνονται υπόψη όλα τα κριτήρια ε, που αφορούν τις επενδύσεις. Σήμερα ή μάλλον το φθινόπωρο, αν πάνω όλα καλά, θα εξεταστεί στην Ολομέλεια αυτή η έκθεση. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει αντιδράσει μετά το δημοψήφισμα της Βρετανίας. Ανάλογα και με το αποτέλεσμα θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε τις 19 χώρες μέλη της Ευρωζώνης, 7 χώρες που ενδέχεται να προσχωρήσουν και 2 χώρες που έχουν opt-out. Πρέπει να δούμε όλους αυτούς τους συσχετισμούς. Κάτι άλλο που δεν πρέπει να μας ε, διαφεύγει είναι ότι έχουμε και την ε, Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων με την έκθεση Μπροκ Μπρέσο που εξετάζει το τι μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της ε, συνθήκης και έχουμε και την έκθεση Φερχόφστατ για το τι μπορεί να γίνει πέραν της συνθήκης. Αυτά ως προς το πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, όπως ο Ράιμερ Μπέγκε, έτσι και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στις απαντήσεις που θα πρέπει να δώσουμε σε τέσσερις ερωτήσεις. Όπως βλέπουμε και από το έγγραφο εργασίας να προκύπτουν. Η πρώτη ερώτηση δεν είναι αν χρειάζεται προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουμε αφήσει πίσω μα αυτό το ερώτημα. Αλλά γιατί χρειάζεται ένα προπολογισμό τη Ευρωζώνη. Γιατί όπω είπα, χωλαίνει αυτή τη στιγμή η ΟΝΕ ναι και πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό. Άρα, τρεις πυλώνες όταν άρχισε να λειτουργεί ο Ευρωπαϊκό Μηχανικός σταθερότητα κάλυψε αυτήν την ανάγκη να απορροφά ασύμετρα σοκ. Αυτό θα πρέπει να το αναλάβει ε, ο νέος προπολογισμό. Δεύτερη λειτουργία του θα ήταν η απορρόφηση των συμμετρικών ε, σοκ και τρίτον σύγκληση εντό Ευρωζώνης. Όλες οι μελέτες από το 8 και μετά δείχνουν ότι αυτό που θεωρεί το δεδομένο, δηλαδή σύγκληση των οικονομιών της Ευρωζώνης, δεν επαληθεύτηκε στην πράξη. Υπήρχαν βέβαια οι όροι του Συμφώνου Σταθερότητας και έγιναν και κάποιες βελτιώσεις μεταξύ των μελών. Δεύτερο ερώτημα. Ποια είναι τα εργαλεία που θα μπορούσαμε να έχουμε στη διάθεσή μας για να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Έχουμε τα κονδύλια δημόσιων ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά σίγουρα χρειάζονται εργαλεία σύγκλησης. Και ενδεχομένως, με βάση τις εργασίες που και εσείς, κύριε Πρόεδρε, έχετε ξεκινήσει όταν η ΣΕΡΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με Φερχόφστατ και Μπρόκ είχατε εξετάσει τον ενδεχόμενο κώδικα δεοντολογίας, ε, κώδικα σύγκλησης μάλλον, για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βγούμε από τα πλαίσια των στον οποίο αυτή τη στιγμή είμαστε περιορισμένοι. και να εφαρμόσουμε τα κριτήρια σύγκλησης. Έχουμε και κάποιες άλλες προτάσεις ε, που είναι πιστικές από οικονομικής πλευράς, ε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε επίπεδο ευρωζώνης να υπάρχει ένας αυτόματος σταθεροποιητής. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι με τους κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης θα μπορούσε αυτό να ξεκινήσει και να γίνει πράξη. Θα μπορούσαμε να έχουμε και να αλλάξει το επίδομα ανεργίας. σε επίπεδο ευρωζώνης. Έχετε και σε επίπεδο Eurogroup και τα λοιπά. Το θέμα είναι πώς μπορεί να εφαρμοστεί από πολιτικής πλευράς. Τρίτο ερώτημα. Οι πηγές χρηματοδότησης για να τροφοδοτηθεί αυτός ο από πού θα προκύψουν. Μαζί με τον Ρέμερ Μπέγκ έχουμε εργαστεί επί του θέματος. Τελικά, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διευκρινιστεί το πώς αυτή η συζήτηση μπορεί να συσχετιστεί με μια άλλη συζήτηση που γίνεται στο Κοινοβούλιο και που αφορά την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αφορά και τα 28 κράτη-μέλη. Αν θέλουμε να έχει αίσιο πέρας η συζήτηση για έναν προπολογισμό της Ευρωζώνης, δεν μπορούμε εύκολα να προεξοφλήσουμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη συζήτηση. Άρα, πρέπει παρότι φυσικά και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα την ύπαρξη τη Ευρωζώνη όταν θα αξιολογούμε ή θα επανεξετάζουμε τον προπολογισμό, το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Τα διαρθρωτικά ταμεία είναι κάτι απαραίτητο. Δεν μπορεί να είναι το α και το ω, ε, αλλά είναι σίγουρα σημαντικά. Και σίγουρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα διαρθρωτικά ταμεία. Βέβαια, ακόμα όλα είναι ανοιχτά, πίστες διαρευνούμε προς το παρόν Μπορούμε να φέρουμε τουλάχιστον τρει. Έχουμε τα ευρωομόλογα από τη μία, βέβαια. Και εδώ δύσκολα τα πράγματα από πολιτικής πλευράς. Ήδη οι πόροι είναι μια δεύτερη δυνατότητα, ειδικοί ήδη οι ποροι ειναι μια δευτερη δυνατοτητα ειδικη ηδη οι ποροι Με την Κεντρική Τράπεζα όταν συζητούσαμε και κατόπιν πρωτοβουλίας ορισμένων συναδέλφων αναφέρθηκε το ενδεχόμενο τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας να μπουν στον προπολογισμό της Ευρωζώνης. Και τέλος, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, από τον οποίο μπορεί να προκύψει μια κρίση μάζα σημαντική για ένα μελλοντικό προπολογισμό της Ευρωζώνης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα ζητούσε να μπει το ESM στην κοινοτική μέθοδο. Είχαμε και την έκθεση των πέντε προέδρων σχετικά, στη δεύτερη φάση το πρόβλεπε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας να δούμε τι περιθώρια θα μπορούσαμε να προτείνουμε για να χρηματοδοτήσουμε το backstop ε, της Τραπεζικής Ένωσης. Ο Ρέμερ Μπέγκε είπε πολλά, δεν θέλω να επανέλθω. Τρία πράγματα θα αναφέρω όμως. Πρώτον, δημοκρατική οικονομική διακυβέρνηση δεν θα υπάρξει αν δεν υπάρξει ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι το Κοινοβούλιο της Ευρωζώνης. Θα πρέπει να διδαχθούμε από το παρελθόν. Στο παρελθόν, όταν δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν όλες οι χώρες μέλη της Ευρωζώνης ή όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ομοφωνίας, επειδή υπήρχε ο κανόνας, έγιναν κάποιες άλλες, μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες άλλες διευθετήσεις, εκτός δηλαδή ε, πλαισίου συνθήκης και η Κομισιόν ε, παίρνει τις πρωτοβουλίες. Ε, έχουμε και το δικαίωμα βέτο, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και λάμβοντας υπόψη και τη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε να επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Δεύτερη πεποίθηση. Μιλούσαμε πάντα για έναν Υπουργό Οικονομικών. Το έχουμε ψηφίσει πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζουμε ότι ταυτόχρονα θα έπρεπε να σκεφτούμε κάτι ενδιάμεσο. Για να πείσουμε αυτούς οι οποίοι από κοινού με εμάς θα μπορούσαν να προωθήσουν την ανάγκη ενός προϋπολογισμού της Ευρωζώνης, μιλώ για τους Υπουργούς Οικονομικών. Και έπειτα έχουμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τι ρόλο μπορεί να έχει. Τελευταίο. Στην Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων, ο συνάδελφος Παύλο Ρανζέλ μελετά αυτή την περίοδο το πώς θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε από το σύστημα του εποπτικού μηχανισμού της Τραπεζικής Ένωσης και να το μεταφέρουμε στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά νομίζω ότι είναι μια σημαντική πηγή έμπνευση που θα πρέπει να την δούμε εκ του σύνεγγυ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Περβάνο Περέ. Θα δώσω το λόγο στου κοιόδη εισηγητέ. Ένα δίλεπτο στη διάθεσή του. Σύγκριτ Μουρεσάνου πρώτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καταρχά, να ευχαριστήσω του δύο συνεισηγητέ για τη δουλειά που έκαναν μέχρι τώρα για τα δύο έγγραφα εργασία που υπέβαλαν και για την ακρόαση που διοργάνωσα τον μήνα Μάρτιο. Το βασικό προς διευκρίνηση είναι γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη δυναμικότητα την φορολογική και την οικονομική. Κατά την άποψή μου, για να βελτιώσουμε την αντοχή των οικονομιών μας εν ώψη νέων κρίσεων. Διότι θα μας πλήξει η κρίση η επόμενη και ξέρουμε πού θα προέλθει. Πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μα για να τα Με ποια εργαλεία. Διαθωτικέ μεταρρυθμίσει. Και υπάρχει στέρεη βάση για τέτοιε μεταρρυθμίσει, Για να δημιουργηθεί αυτό το οικονομικό δυναμικό στην έκθεση των τεσσάρων προέδρων. Συμφωνώ στι ηγητές. Πρέπει να αξιολογήσουμε τα διαθέσιμα εργαλεία. Πιστεύω βασικό εργαλείο προς εξέταση είναι η συστάση κατά χώρα. Βλέποντα αυτέ, βλέπουμε ότι αυτό πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Όλοι όμως απογοητευόμεθα διότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται. Αν καταφέρουμε οικονομικά να δώσουμε κίνητρα για τις χώρες, για τις καταχώρες συστάσεις, αυτό είναι το σωστό εργαλείο για να ελοποιηθούν. Σχέση μεταξύ Ευρωζώνης και μη Ευρωζώνης. Έχουμε 19 κάτι μέλη της Ευρωζώνης. Τα κράτη-μέλη εκτός Ευρωζώνης δεν έχουν υποχρέωση να προσχωρήσουν μόνο δύο. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία. Οι χώρες εκτός Ευρωζώνης που μεσοπρόθεσμα θα ενταχθούν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν στις οικονομικές δυνατότητες όσον αφορά συνεισφορές, τα ευεργετήματα και η διακυβέρνηση. Τέλος, πρέπει να είμαστε πραγματιστές όσον αφορά το οικονομικό δυναμικό που θα δημιουργήσουμε. Τι είναι πολιτικώ εφικτό να μην κάνουμε και εμείς αυτά που να κάνουν οι άλλοι. Το ESM ε απο, απορροφά τους κλειδονισμούς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η τελευταία γραμμή άμυνας. Ζητά ο Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας να κάνουν πράγματα οι Υπουργοί Οικονομικών σε κράτη-μέλη, να κάνουν μεταρρυθμίσει, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών του και να γίνουν ανθεκτικέ οικονομίε έναντι τη επόμενη κρίση. Ευχαριστώ. Ο Πολ Τόγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εισηγητές για την έρευνα που έκαναν και για τα έγγραφα. Και εγώ ανησυχώ όπως και ο Χάιμα Μπέργκα Και με τι ανησυχίε του πρώτη. Επικίνδυνη είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε ένα κοινό νόμισμα. Αλλά δεν έχουμε κοινή πολιτική. Διότι δεν έχουμε κοινά εργαλεία. Άρα, κάποτε υπάρχει πιθανότητα η Ευρωζώνη να καταρρεύσει και να διαλυθεί και να διασκορπιστεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν να πρέπει να προετοιμαστούμε την επόμενη κρίση στα πλαίσια των πολιτικών περιορισμών. Τι θα γίνει αν ε, ε, αποτελματωθεί η Ευρωζώνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποια θα είναι η ανταπόκριση. Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά που κάνουμε είναι μια προετοιμασία για την επόμενη κρίση. Άρα, χρειαζόμαστε μια τραπεζική ένωση που πρέπει να ολοκληρωθεί και να σπάσει ο κρίκος μεταξύ κρατών μελών και τραπεζών. Κρίσιμο αυτό. Επίσης, να υπάρχει δυναμικό απόθεμα, ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν σταθεροποιητικές πολιτικές. Χωρές αυτές, κλειδονισμοί συμμετρικοί και ασύμμετροι θα πλήξουν την ευρωπαϊκή οικονομία και πολύ και δεν θα έχουμε επαρκή απάντηση. Λοιπόν, ε, ε, σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει πρόβλημα ε, ανταπόκριση στα οικονομικά προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλο χρέο. Δεν μου αρέσει ο τίτλο τη εκθέσεω, αναφέρεται στο εργαλείο. Πρέπει να θέσουμε του στόχου. Να προτάξουμε του στόχου. Η βάση τη Ευρωζώνη, τα θεμελιώδη προβλήματα τη Ευρωζώνη, πώ θα σταθεροποιείται ε, η Ευρωζώνη μέσω των καταλήλων πολιτικών. Τούτου λεχθέντο. Οι συγητές προσπαθούν να βρουν διεξόδους για τα καινούργια εργαλεία εντός του δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Αυτό είναι κρισίμου σημασία. Διότι έτσι θα έχουμε ελεγκτικό μηχανισμό και μηχανισμό διακυβέρνησης δημοκρατικά στοιχεία. Και στην Ευρώπη λείπει ο δημοκρατικός έλεγχος και δημιουργείται ε, η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι τεχνοκρατικό και έχει πολιτικό, αλλά είναι πολιτικό. θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίε των δύο επιτροπών, της Επιτροπής Προπολογισμών και Οικονομικών. Για να μην φαίνεται ότι τα κάτι μέλη εκμεταλλεύονται ε, τα, τις οικονομικές πτυχές της προσπάθειας χωρίς να κάνουν προσπάθεια για την κοινή προσέγγιση σε όλα τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Κύριο Σκορμπέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους ε, δύο εισηγητές για τη δουλειά που έχουν κάνει και θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για προϋπολογισμό της Ευρωζώνης να θυμόμαστε το πρώτο κομμάτι που λέει Ευρωζώνη. Τι είναι το ευρώ? Το ευρώ σημαίνει ως κοινό νόμισμα ότι τα κράτη-μέλη της ΟΝΕ δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να διορθώσουν τα προβλήματα της οικονομίας τους μέσω της προσαρμογής της ισοτιμίας. Αυτό είναι θεμελιώδες πρόβλημα και το γνωρίζαμε πάντα, αλλά υπήρχε κάποια ελπίδα ότι η ανταγωνιστικότητα θα προσαρμοζόταν συν το χρόνο. Και άρα δεν θα ήταν αναγκαία η προσαρμογή μέσω των νομισματικών ισοτιμιών. Το 2016 βεβαίως είμαστε στο 8ο έτος κρίσεως και όποιος λοιπόν λέει ότι το ευρώ θα μας οδηγήσει σε κάποιον παράδεισο ανταγωνιστικότητας, προφανώς δεν βλέπει την πραγματικότητα. Είτε θα αντιδρούσαν όλοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν το κάνουν, οπότε χρειάζονται κάποιες διαφορές. Και οι χώρες οι οποίες δεν μπορούν εδώ πέρα να ακολουθήσουν, θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αποχωρήσουν. Και άρα εδώ πέρα δεν βλέπω πώς μπορούμε να μιλάμε για προπολογισμό της Ευρωζώνης χωρίς να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Ε, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Π.χ. πώς μπορούμε να εξηγήσουμε σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βγαίνουν οι πολίτες ε, στα 58 ή στα 60 στην σύνταξη, ενώ άλλοι σε άλλες χώρες θα βγαίνουν σύνταξη στα 67 ή στα 70 λέμε τώρα. Δηλαδή μπορούμε να το λέμε, αλλά το θέμα είναι υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες εξισωτικές πληρωμές και αν ναι, από πού προκύπτουν. Ουσιαστικά η Ευρωζώνη θα γίνει μια ένωση δημοσιονομικών μεταβάσεων η οποία δεν είχε προβλεφθεί ποτέ. Και τελευταία σκέψη. Έχουμε την συνθήκη του Μάστριχτ και δικαίω είπε ο κύριος ε, Μπέγε ότι θα πρέπει να τηρούμε τις συνθήκες. Μα δεν τηρούμε τη συνθήκη του Μάστριχτ. Εκεί πέρα ορίζεται ξεκάθαρα 3% ετήσιο χρέος το έτος, 60% ανώτατο όριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι καλό που βλέπουμε ότι στο πάνελ των εμπειρογνωμόνων που ακούσαμε πρόσφατα ανελήφθη, αναφέρθηκε ο κίνδυνος, ο ηθικός κίνδυνος. Εάν υπάρξουν ανεξέλεκτες μεταφορές οικονομικές Θέλουμε λοιπόν να ελέγχονται κάπως οι πολιτικές των κρατών μελών και όπως είπε το πάνελ, μέχρι τώρα οι εμπειρίες δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Δείχνουν ότι δεν υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες συντονισμού. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ελέγξουμε τα διάφορα ηθικά προβλήματα, του ηθικούς κινδύνους, αλλά είναι μικρές οι δυνατότητες. Συζητούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το καταλάβουμε να κατευθύνουμε τι πολιτικέ των κρατών μελών. Είναι τεράστια μετακύληση κυριαρχία από τα κράτη-μέλη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα είναι άχρηστα όμω τα δημοκρατικά συστήματα των κρατών μελών να γίνει αυτή η μετακύληση, αυτή η μεταφορά. Δεν λέμε αν θα είναι κάτι εφικτό ή επιθυμητό όσον αφορά τη δημοκρατία και τον προπολογισμό και τη χρηματοδότησή του. Στο έγγραφο εργασία που συζητούσαμε με του συναδέλφου, αναφέραμε τη χρήση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ο μηχανισμός σταθερότητας όμως είναι μηχανισμός διαχειρίσεως κρίσεων και μέτοχοι είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποφασίσει μόνη της για τη χρήση αυτού του ποσού. Το ίδιο αφορά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα χρήματα μοιράζονται στις Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες που ελέγχουν και είναι ιδιοκτήτες Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να επιθυμούν τα κράτη-μέλη μπορούν να προκαταβάλουν τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Ίσως τα προβλήματα ε, οφείλονται στη διοικητική δομή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, περιέχονται ανισορροπίες. Χρειάζεται το σωστό κράμα πολιτικών. Θα μεταφέρονται τα κράτη-μέλη εθνικοί πόροι προς μία δομή κυβερνητική όπου όλοι θα πρέπει από κοινού να αποφασίζουν για τη χρήση των χρημάτων. Ένα είδος θησαυροφυλάκιο για την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση θα ήταν. Αυτό αφορά μια συζήτηση περί δημοκρατικής νομιμότητας. Μάλλον δύσκολο να το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Καμιά φορά είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς την πραγματικότητα, γιατί συνήθως νικάει η πραγματικότητα. Όμως προσβλέπω σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση επί του θέματος αυτού και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον Ρέμερ Μπέργκερ και τη Μαρβάν Σμπερέζ για τη δουλειά, την αξιοσημείωτη που πετέλεσαν. Η Ευρωζώνη από ό,τι φαίνεται πιθανότατα κινδυνεύει σήμερα. Όταν θεσπίσαμε το ενίο νόμισμα, διερωτηθήκαμε χρειαζόταν οικονομική διακυβέρνηση ή απαιτεί το κάποιος κανόνας ε, συνειδιοκτησίας, κανόνες συνειδιοκτησίας που θα καθόριζαν κριτήρια προς ε, συμμόρφωση των κρατών μελών εκείνων που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το νόμισμα. Η επιλογή έγινε, επιλέξαμε τον κανονισμό χωρίς την οικονομική διακυβέρνηση, τι διαπιστώνουμε σήμερα, ότι ο κανόνας δεν γίνεται πλέον σεβαστός έχουν γίνει πολλές παραβάσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, δεν υπάρχουν πλέον κανόνες και δεν υπάρχει και διακυβέρνηση. Κυβέρνηση. Δεν υπάρχει οικονομική πολιτική στην Ευρωζώνη. Κάθε κάτος μέλος υλοποιεί τη δική του οικονομική πολιτική. Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας για το Ευρωκοινοβούλιο αποτελεί μια ευκαιρία. Ευκαιρία να μιλήσουμε στους Ευρωπαίους και να προβούμε σε μια διδασκαλική προσπάθεια παιδαγωγική προσπάθεια. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Θα ήθελα λοιπόν η συγητής να κάνει την επιλογή της τόλμης στην πρόταση που θα γίνει. Να μας προτείνουν οι συγητές το βέλτιστο σχήμα ώστε η Ευρωζώνη να είναι μια οικονομική ε, ζώνη βέλτιστη. Είναι αυτό που συνάδει με τις παρούσες συνθήκες. Υπάρχουν και κάποιες απαιτήσεις προς τροποποίηση των συνθήκων. Ε, θα πρέπει να έχουμε φιλοδοξία, να προτείνουμε το ιδέωδες σχήμα προς το οποίο θα πρέπει να κινηθούμε ώστε επιτέλους οι ευρωπαϊκές υποσχέσεις ε, να υλοποιηθούν. Διότι, προσέξτε το εξή. σε πολλές περιστάσεις κάθε φορά ανακοινώναμε σημαντικές προόδους όσον αφορά την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όμως πολλαπλασιάσαμε τις απογοητεύσεις και τις αποτυχίες. Και βλέπουμε σήμερα την άνοδο του λαϊκισμού Οπότε κατεπηγόντως πρέπει να κινηθούμε. Καλό τους ηγητές που έκαναν πολύ καλές προσπάθειες να αποδειχτούν τολμηροί. Υπάρχει πάντα χρόνος να βρούμε το μονοπάτι του εφικτού. Πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, την εκπαιδευτική. Σας εμπιστεύω, ευχαριστώ Ζαν, για την έκκλησή σου για φιλοδοξία. Ο Νίλς Τόρβαλς. Νίλ δεν είναι εδώ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω εκ μέρους του. Θα μιλήσω γαλλιστή, ακόμα και ο Νίλσε θα μιλούσε γαλλικά βέβαια. Καταρχάς ευχαριστούμε για τη δουλειά που είναι αξιοσημείωτη. Δεύτερον πιστεύω ότι ο Ζαν Αχτουή το είπε και ο κύριος Τάγκ. Ο πραγματικός λόγος της προσπαθίας και της εργασίας είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλή ανεργία και ελάχιστη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να περάσουμε από πανεπιστημιακές εκθέσεις, θεωρητικές εκθέσεις στη δράση, όπως λέει η κυρία Μπερές. Όχι για να ικανοποιηθούμε ή να αλλάξουμε τους θεσμούς, αλλά διότι υπάρχει πραγματική ανάγκη. Δεύτερον, θεωρώ ότι μπορούμε να αναπτύξουμε την έννοια του δημοσίου αγαθού. Όταν πολιτική οντότης δημιουργείται, ε, δημιουργούμε έναν προϋπολογισμό για χρηματοδότηση. Είχαμε πάλι σαν έναν του στόχου την νομισματική σταθερότητα κλπ. Δημιουργήσαμε διάφορου θεσμού για αυτόν τον σκοπό. Η αναθεώρηση των συνθήκων είναι το τρίτο σημείο. Παρόλο που επικρατεί πλήρη σύγχυση, βρίσκεται στη ρύθμιση που επετέχθη για το Ηνωμένο Βασίλειο, το settlement. Δεν ξέρω ποια είναι η νομική υπόσταση της πράξης, η υλοποίηση θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα πιθανότατα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αορίστως κάπου υπόσχεση αλλαγή των συνθήκων. Θα πρέπει λοιπόν να ενταχθούν σε αυτή την προοπτική. Αν βγει το Ηνωμένο Βασίλειο, όμως τότε δημιουργούνται άλλες προοπτικές, αλλά πιθανότατα πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες της συμβιώσεώς μας θα επέμενα επί ενό σημείου που θεωρώ σημαντικότατο του πολίτε, δηλαδή σαφήνεια, σαφήνεια των δικαιωμάτων και των ευθυνών. Δεν μπορούμε πλέον να λειτουργήσουμε σε ένα σύστημα στο οποίο ζήσαμε επί του προσωρινού. Κατανοούμε ότι το Μάστριχτ ήταν προσωρινό. Θεωρούσαμε ότι τα κάτι μέλη θα έμπαιναν στην Ευρωζώνη. Αυτό ανεφερόταν επί χάρτου στο πρωτόκολλο υπαριθμών 12. Αλλά επειδή θεωρούσαμε ότι είχαμε, ακροπόθεσμα θα έμπαιναν όλοι, είχαμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο εκεί και το σέτλουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά, η ρύθμιση αυτή του Ηνωμένου Βασίλειου για πρώτη φορά μετά τη δημιουργία του νομίσματος, υπονοεί ότι δεν υπάρχει μόνο ένα νόμισμα της Οικονομικής Νομισματικής Ενώσεως, που είναι το νόμισμα της Ενώσεως, που είναι το ευρώ. Είχαμε ένα νέο πλαίσιο για ένα νέο νόμισμα. Αν, δεν έχουμε, αν έχουν πολλά νομίσματα, δεν υπάρχει λόγος για νέο πλαίσιο. Νομίζω ότι από αυτού πρέπει να είμαστε σαφέστατοι. Όλες οι άλλες λύσεις που να λέμε ότι είναι κάποιοι που είναι μέσα λίγο απ' έξω και παίρνουν αυτό που τους ρυθμίζει αυτά δεν μπορούμε να τα ανεχθούμε και να τα προβάλλουμε στους πολίτες όλοι είναι πρόσδεκτοι στην Ευρωζώνη όλοι αυτοί που είναι έτοιμοι να υπομισθούν τις ευθύνες όλες έχουν όλα τα δικαιώματα εκείνοι που δεν λαμβάνουν τις ευθύνες που δεν, δεν είναι μέλη του νομίσματος και λοιπόν δεν έχουν καμία σχέση με τα αποφασιστικά τα όργανα λήψης αποφάσεων αν δεν το ξεκαθαρίσουμε αυτό ότι πρέπει να εφεύρουμε κάτι άλλο από αυτό που είχαμε μέχρι τώρα Νομίζω ότι τότε θα διαιωνίζουμε ένα περίπλοκο χαρακτήρα των πραγμάτων που δεν είναι κάτι δύσληπτο για τους πολίτες και δημιουργεί πραγματικά προβλήματα όσον αφορά τη δημοκρατία. Προσωπικώ πώ πιστεύω ότι ο προπολογισμό Ευρωζώνη κάποια στιγμή σημαίνει ένα κοινοβούλιο τη Ευρωζώνη. Πίσω εντό του κοινοβουλίου να υπάρχουν επικαλύψει χωρί να υπάρχουν επικαλύψει, όσο αποκλείεται κανεί, μπορεί να συμμετέχει στι συζητήσει. Αλλά τη στιγμή θα ψηφίζουμε, που ελέγχουμε τι εκτελεστικέ αρχέ, τι ημέρε που αποφασίζουμε για τη χρήση των χρημάτων, τα μέλη τη Ευρωζώνη θα είναι εκείνα που θα αποφασίζουν. Και ό,τι είναι περίπλοκο, κάποια δεδομένη στιγμή θα καταλήξει να στραφεί εναντίον μα. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συνεισηγητές και εγώ. Για... Κοιτάξτε, για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένα κοινό μέσο για να αντιμετωπίσουμε τι μελλοντικέ κρίσει, πρέπει να εστιάσουμε σε πολλού τομεί κλειδιά. Ακριβώ για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και την έλλειψη ανάπτυξη και όπω ήδη αναφέρθηκε και στην ε, λογική της ε, ανάπτυξης ε, των δημοσίων αγαθών θα θέλαμε να σκεφτούν οι εισηγητές τα εξή θεωρώ πως πρέπει να υπάρξει ένας χρυσός κανόνας επενδύσεων καθώς οι επενδύσεις δημιουργούν έσοδα και για τις μελλοντικέ γενναίες. Και βεβαίως με τις, ε, οι δημόσιες αυτές επενδύσεις θα πρέπει να εξαιρούνται από τους ε, κανόνες χρέους ε, και ελλείμματος του Συμφώνου Σταθερότητας. Οι δυνατότητες αυτές μέσω των επενδυτικών τραπεζών της Ευρώπης, μέσω διαφόρων εγγύσεων, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ερευνήσουμε. Έτσι θα συμπληρωθεί η νομισματική πολιτική, η οποία αυτή τη στιγμή κολλάει λόγω της δημοσιονομικής λιτότητας και δεν μπορεί έτσι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ανταποκριθεί στην εντολή της. Τέλος, χρειαζόμαστε περισσότερες ε, συνεισφορές ε, από τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλες ανάλογες τράπεζες και στις δημόσιες τράπεζες για να προωθηθούν οι επενδύσεις οι οποίες θα πρέπει να εξαιρούνται από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δεν βλέπω τον Φάμπιο μαζί. Υπάρχει άλλος ένας ομιλητής ε, για την Κουένε, Έρνεστ Μαργκάλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πλήρες το έγγραφο, είναι άρτιο και νομίζω ότι γύρει θετικές προσδοκίες. Όμως υπάρχει και ένας κίνδυνος να γίνουμε αυτάρισκοι ή ως κοινοβούλιο να στείλουμε ένα με μεν ε, μήνυμα εφόσον ορίζουμε πολύ σωστά τον χαρακτήρα και τις δυνατότητες αυτές τις δημοσιονομικές για την Ευρωζώνη, για τους στόχους, για τις λειτουργίες, κίνδυνους, κινδύνους ευκαιρίες κτλ, κτλ. Όλα αυτά τα έχουμε εντάξει, όμως. Η έκθεση αυτή θα κρυθεί σε σχέση με τον πραγματικό αντίκτυπο που θα έχει. Και όχι με το τι λέει απλά και το που εστιάζει. Αν μπορεί να χαρακτηριστεί μάλιστα υποθετικό για να μην πω ουτοπικό το περιεχόμενό της. Το θέμα είναι δηλαδή στην πράξη. Αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι με την Κομισιόν και το Συμβούλιο που είναι και απαραίτητο αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Επίσης, άλλος κίνδυνος να δεχθούμε ότι η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύο έννοιε που θα συμβιώνουν εκ παραλίλου, για πάντα σχεδόν. Δημοσιονομική ικανότητα, τι σημαίνει. Σταθεροποίηση, ικανότητα για δικαιωτικές πολιτικές, επενδύσεις, το έχω ξαναπεί. Σημαίνει επίσης αναδιανεμητική δυνατότητα και καθορισμός των πολιτικών με βάση την παροχή κοινοφελών υπηρεσιών και υπηρεσιών ε, δημοσίου συμφέροντος και ενδιαφέροντος. Πρέπει να δούμε όμως πώς θα περάσουμε από ένα μηχανισμό μόνιμων ε, μεταφορών πιστώσεων όπως μέχρι τώρα σε μια συνυπεύθυνη αλλαγή ενώ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που μας ενημερώνει για τις ανισορροπίες. Αυτό είναι η μία κατεύθυνση. Θα πρέπει να δούμε όμως και τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα και να αντιμετωπίσουμε με την ίδια λογική και να υπάρχει δυνατότητα επιβολή κυρώσεων και για τις δύο περιπτώσεις, όχι μόνο για τα ελλείμματα. Ναι, ναι, ναι. Τι έπρεπε να... Είχα δύο λεπτά α, μόλι, μόνο. Έχουμε και το μηχανισμό σταθερότητα, αλλά αυτός πρέπει να είναι η βάση για τη δημιουργία ε, και μια πραγματική ενό επενδυτικού, ταμείου επενδυτικού προγράμματο. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για το έγγραφο εργασίας που μέχρι στιγμής τουλάχιστον θέτει τα σωστά ερωτήματα και τώρα είναι ώρα να πάρουμε και τις σωστές απαντήσεις πιστεύω. Όπως όλοι πιστεύω έχουν τονίσει και εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και γνωρίζουμε ότι δεν μας αντιμετωπίζουν όλοι ως ένα καταπληκτικό θεσμικό όργανο, γιατί όλοι νομίζουν ότι θέλουμε όλο και περισσότερα ε, χρήματα, όλο και περισσότερα κτλ. κτλ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί δηλαδή θέλουμε να υπάρχει αυτή η δημοσιονομική ικανότητα. Και η απάντηση είναι ότι θέλουμε να εξομαλύνουμε τα ασύμετρα σοκ. Αυτό είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο συζητούμε και θέλουμε να περάσει αυτή η πρόταση. Και ήδη και από τον τίτλο θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν συζητούμε έτσι και μόνο γιατί μας αρέσει να συζητάμε αυτό το εργαλείο, αλλά το πρόβλημα της Ευρωζώνης, όπως έχει αυτή τη στιγμή, είναι ότι χρειάζονται περισσότερα εργαλεία, διότι το είδαμε και στην προηγούμενη κρίση, ότι έπρεπε να δημιουργηθούν μέτρα και να εφαλοποιηθούν μέτρα κατεπήγοντα στα οποία ασκήθηκε έντονη κριτική. Αλλά αυτό έγινε γιατί δεν είχαμε επαρκή εργαλεία. Και αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε τώρα. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Και εξηγεί και γιατί έχουμε αυτή τη συζήτηση. Τώρα έρχομαι ε, στο πλαίσιο και έχω κάποιε ερωτήσει προ του εισηγητέ. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε έναν ημιαυτόματο σταθεροποιητή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν συμφωνούν να δημιουργηθούν όλες αυτές οι αιρεσιμότητες γιατί είναι σημαντικό να υπάρξει μεγαλύτερη αυτοματοποίηση, αυτοματισμό. Αν θέλουμε να έχουμε πολιτικέ συζητήσει για τι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει κτλ., μπορούμε και το κάνουμε ούτω ή άλλω. Έχουμε το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη και να σα πω ότι και το ελεγκτικό συνέδριο λέει ότι πρέπει αυτά τα εργαλεία να βελτιωθούν. Α μην επιβάλλουμε αυτή τη συζήτηση όμω ε, στην ε, σημερινή συζήτηση για του ε, σταθεροποιητέ τώρα. Πέρασε ο χρόνο μου από ό,τι βλέπω, αλλά για να ολοκληρώσω. Κάτι ακόμη σημαντικό είναι η ηθική κίνδυνη και οι μόνιμες και τα λοιπά. Αν δημιουργηθεί ή αν είχε δημιουργηθεί όταν δημιουργήθηκε και η Ευρωζώνη ένα αντίστοιχο εργαλείο, η Γερμανία κατά πάσα πιθανότητα θα είχε επωφεληθεί από αυτόν τον αυτόματο σταθεροποιητή και θα είχε αποφευθεί η φούσκα στην Ισπανία που ήταν ένα από τα προβλήματα ε, της κρίσης. Άρα θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι ένας τέτοιο σταθεροποιητής δεν σημαίνει ότι θα έχουμε μόνες φορέ πιστώσεων από το βορρά προς τον νότο, αλλά ότι θα είχε βοηθήσει στο παρελθόν πολλέ χώρες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους αυτό ο σταθεροποιητή. Και αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να μεταπίσει και αρκετού και να ταχθούν υπέρ. Μάρκο Τζάνι τώρα. Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ τους δύο συνηγητές για την πολύ λεπτομερή εργασία που έκαναν προετοιμάζοντας τα δύο έγγραφα. Δυστυχώς αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αυτή η συζήτηση είναι άλλη μια μάταιη προσπάθεια διάσωσης ενός ασθενούς που τώρα πλέον έχει αποθάνει η Ευρωζώνη και μετά θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί. Είναι ένα εγχείρημα που οικονομικά και πολιτικός είναι ε, μη βιώσιμο και η συζήτηση για τον προπολογισμό της Ευρωζώνης ε, το αποδεικνύει αυτό. Από αυτά που γράφουν και τα έγγραφα το βλέπουμε και, και κάποιες ε, συνέπειες που υπάρχουν μεταξύ εκείνου που απαιτείται και θα χρειαζόταν ούτω ώστε να λειτουργεί η Ευρωζώνη και να είναι βιώσιμη και εκείνου που είναι πολιτικός αποδεκτό. Όποιος διάβασε τις εργασίες του Ρόμπερ Μούντερ γνωρίζει ότι για να υπάρχει μια τέτοια βέλτιστη οικονομική ένωση που λειτουργεί, όπως δεν είναι σήμερα Ευρωζώνη, απαιτούνται κάποιες ε, ρυθμίσεις, κάποια εργαλεία. Και εδώ ξεκινάνε οι συνέπειε στο έγγραφο, στα έγγραφα που συνετάχθησαν γίνεται λόγος προφανώς για τη δημιουργία ενός εργαλείου που δεν γίνεται ένα εργαλείο μεταφοράς μόνο μερούς μόνιμης. Όμως δυστυχώς αυτό χρειάζεται για να καταστεί λειτουργική ευρωζώνη, δηλαδή ένα εργαλείο μεταφοράς μόνιμης οικονομικής και φορολογής από τις, από χώρες που πιστώνουν προς εκείνες που είναι χρεωμένες. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Η διασύνδεση του προπολογισμού της Ευρωζώνης με τις διαθετικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να θεσμοθετηθεί, να θεσμοποιηθεί η Τρόικα και εκεί υπάρχει πρόβλημα δημοκρατικού ελέγχου. Το βασικό και το πιο κρίσιμο σημείο είναι ότι η κατάσταση είναι πολιτικά μη βιώσιμη. Διότι όπως σε μια κρόαση που διεργανώσουν πριν από δύο εβδομάδες περίπου στο Ευρωκοινοβούλιο, ο καθηγητής Απίρ εξήγησε ότι για να καταστεί αποτελεσματικό αυτό το μέσο, αυτό το εργαλείο, χώρες όπως η Γερμανία θα πρέπει να δεχτούν, να θέσουν επιτάπητος, να μεταφέρουν 2,3 ε, ε, ευρώ το χρόνο προς την περιφέρεια. Λοιπόν, ρωτά τους Γερμανούς συναδέλφους πώς θα εξηγήσουν αυτοί στους εκλογείς τους ότι για να διατηρηθούν οι χώρες που χρωστούν θα πρέπει να ξοδεύουν 200 με 300 δις ευρώ. Αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να βρεθεί απάντηση. Ευχαριστώ Μάρκο Βάλλη, ευχαριστώ Πρόεδρε πέρα από τον συνάδελφό μου και ένα άλλο μέλος του ECR ε, δεν άκουσα κανέναν εστιάζεται σοβαρά επί του προβλήματος της Ευρωζώνης ή του ενιαίου Ένα νόμισμα που δεν ε, κατάφερε να είναι το νόμισμα 19 χωρών, δεν θα είναι για 28, έφερε μόνο κλειδονισμούς, ανισότητες, ανισορροπίες, ανισορροπίες όπου οι χώρες που έχουν πλεόνασμα πρέπει να πληρώνουν ή να στηρίζουν τις χώρες που έχουν έλλειμμα όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο και έχουμε αυτή την ανισορροπία και τα κριτήρια της ε, σύγκλησης για τη βέλτιστη οικονομική ζώνη ε, ποτέ δεν θα εφαρμοστούν διότι ένα πολιτικό πρόβλημα δημιουργείται με αυτή την προσέγγιση ένας προπολογισμός με ρησιμότητες οδηγήσει σε άλλη μια καταστροφή. Είδαμε ότι αν θέτεις κανόνες και ρησιμότητες ε, για ποιους ισχύουν, ε, για κάποιες χώρες ισχύουν, για άλλες όχι και δημιουργείται ένας μηχανισμός και μετά δεν ισχύουν οι κανόνες και δεν γίνονται σεβαστοί. Διερωτώ με λοιπόν για να, τι να ξαναπροτείνουμε τέτοιο σύστημα που θα πρέπει να λειτουργεί με τον τρόπο. Μετά η λαϊκή εντολή λείπει. Κανείς δεν συζητά εδώ, σε αυτή την έδρα, το γεγονός ότι αποφασίζουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο framework. Αναφέρεται στην έκθεση των πέντε προέδρων αυτό και σε διάφορα κείμενα, όμως ποτέ δεν ζητήθηκε από τον κόσμο ποια είναι η άποψή τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, να αναθέτουμε στους τεχνοκράτες όπως είναι ο Μόντι και άλλοι και να μην ακούμε τον κόσμο, το λαό. Αυτό θα οδηγήσει σε προβλήματα και κατάρρευση την Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναθεώρηση των συνθήκων είναι κάτι που αναφέρεται. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ενταχθεί μια ρήτρα δηλαδή τη δυνατότητα Οπτά ότι μια χώρα που αποφασίζει δημοκρατικώ μέσω ε, λαϊκού δημοσιοφίσματο ότι θέλει να βγει προ την έξοδο του ευρώ για να σωθεί η χώρα και να ακολουθηθεί άλλο πολιτικό πρόγραμμα διαφορετικό από αυτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με το πολιτικό πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση το, επιβάλλουν ε, οι ομάδε πίεση και όχι οι πολιτικοί. Είναι σημαντικό λοιπόν να θεσπιστεί αυτή η δυνατότητα μια κυβέρνηση που δημοκρατικά έχει εκλεγεί, αν θέλει να αλλάξει κατεύθυνση σε σχέση με αυτή που επιβάλλεται από τα λόμπι και από την ε, Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω το συνάδελφο του ΙΕΝΕΦ η Σοφή Μοντέλ, Χάινεμανς, κύριος Χάινεμανς, όχι. Καλώς. Πάμε στη διαδικασία του Catch Ο κύριος Λεβαντόφσκι είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ. Είναι τίμιο το έγγραφο των συνεισηγητών. Δεν είναι ευσεβής πόθη, αλλά παρουσιάζει ρεαλιστικά την κατάσταση. Μετά από αρκετά χρόνια συζητήσεων μιας μουσουλμικής δυνατότητα για την Ευρωζώνη, μετά όμως από όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς δεν έχουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις. Η κυβερνητική λογική για τη διάσωση του ευρώ φαίνεται να υπερτερεί ως κοινοτική λογική και σε ό,τι ε, βλέπουμε να γίνονται κάποια πράγματα στα, στον τομέα των εσόδων. Αλλά έχουμε και ε, σίγουρα ε, την εχθρότητα των πολιτών απέναντι στους νέους φόρους και τα λοιπά έχουν προτάσεις ομάδος Μόντι. Αν έχουμε τώρα ε, τη δανειοδότηση μέσω του ESM, σημαίνει ότι πρόκειται για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μετά έχουμε το EFSI που χρηματοδοτεί τις επενδύσεις. Έχουμε ε, άλλους μηχανισμούς, επίσης ανάλογα με την περίπτωση. Είναι σαν να δίνουμε καρότα τι για μαστίγιο. Αλλά αυτό το καρότο έχει και ηθικούς κινδύνους. Μία χώρα που δεν είναι ακόμα στην Ευρωζώνη, αλλά είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται λόγω συνθήκης να ενταχθεί κάποια στιγμή. Όμως, είναι αποθαρρυντικά όλα αυτά που προτείνονται. Παραδείγματο χάρη νέα φορολογία, το νέο ομοσπονδιακό μοντέλο. Γιατί αυτή η ιδέα για την απορρόφηση των ΣΟΚ έχει κάποια φεντεραλιστικά στοιχεία. Οι πόροι δεν είναι ε, άπειροι και όλα αυτά που γίνονται γίνονται σε βάρος του προπολισμού όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κύριε Ντανούτα Χούμπνερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε τη συζήτηση για τη δημοσιονομική δυνατότητα από την εμβάθυνση της ε, δημοσιονομικής ολοκλήρωσης της ΟΝΕ. Αυτό θεωρώ πως αυτές οι συζητήσεις ε, θα πρέπει να αφορούν και την μεταρρύθμιση στην διακυβέρνηση της ΟΝΕ. Δεύτερον, θεωρώ πως έχουν γίνει πολλά πράγματα για να προετοιμάσουμε το έδαφος για μια πραγματικά νέα δημοσιονομική δυνατότητα της ΟΝΕ. Υπάρχουν και συνταγματικοί κανόνες, δημοσιονομικοί έναν ισχυρό μηχανισμό οικονομικής βοήθειας, ε, δανεισμού. Νομίζω λοιπόν πως έχουμε προχωρήσει όσον αφορά την ενίσχυση του προϋπολογισμού. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι η σύγκληση σήμερα απαιτεί πολύ λιγότερα όσον αφορά τις επενδύσεις σε σχέση με 15-20 χρόνια. Τώρα, για τη χρηματοδότηση αντιλαμβάνομαι, θα το δω βεβαίω, ελέγχεται αυτό που λέω, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι πάμε πέρα από τους γενικούς κανόνες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και βεβαίως παραβιάζεται η αρχή του ενιαίου προϋπολογισμού και πάμε σε διακυβερνητικέ συμφωνίες. Νομίζω λοιπόν πως καλύτερα είναι να μείνουμε στον προϋπολογισμό που έχουμε, τον ενιαίο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει προσέγγιση η οποία θα βασίζεται σε κάποια κίνητρα και όχι αντικίνητρα και κυρώσεις. Ευχαριστώ. Αλένα Μασούρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στους ε, εισηγητές. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμη η δουλειά μας. Αν μας βοηθήσει να ξαναπατήσουμε στη γη, να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε και να διαλύσουμε τις αμφισημίες που στρέφονται γύρω από την έννοια του προϋπολογισμού της Ευρωζώνης. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι πολιτικές, οι μεγάλες πολιτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε από πλευράς κρατών μελών για τη χρηματοδότηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα εξαφάνιζαν ως διαμαγείας όταν αφορά τις χώρες Ευρωζώνης. Αν θέλουμε να δημιουργηθεί προϋπολογισμός της Ευρωζώνης, όπως είπαν διάφοροι μιλητές και συγκητές, θα πρέπει να το δικαιολογήσουμε από τη χρηματοδότηση πολιτικών ειδικών για την Ευρωζώνη που δεν θα ισχύουν για τα άλλα κράτη-μέλη. Τα... Κάτι το οποίο δεν βλέπω. Εκτός αν επανεφεύρουμε τα διαθωτικά ταμεία με μια πολιτική αιρεσιμότητα. Παρομοίως δεν κατανοώ πώς οι πολιτικέ δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε τον κανονικό προπολογισμό θα εξαφανιστούν για τον προπολογισμό τη Ευρωζώνη, γιατί η κυβέρνηση. Δεν είναι ότι επειδή δίνουμε τον τίτλο του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομία σε μια προσωπικότητα ότι θα έχει μεγαλύτερη εξουσία και μεγαλύτερη επιρροή από ότι έχει ύπατη εκπρόσωπος παραδείγματος χάρη για την εξωτερική πολιτική όσον αφορά τους ίδιου πόρου. δεν κατανοώ πώς τα κάτι μέλη που συστηματικά αντετάχθησαν στην δημοσιονομική αλληλεγγύη για να βοηθήσουν τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, την κρίση Ευρωζώνης ξαφνικά θα δεχόταν τη δημιουργία ε, νέων πόρων για τη χρηματοδότηση νέου προπολογισμού. Νομίζω ότι η ιδιαιτερότητα της Ευρωζώνης ποια είναι, ότι εντός Ευρωζώνης χρειαζόμαστε πραγματική νομισματική και χρηματοστητική αλληλεγγύη, αυτό γίνεται μέσω μεταρρυθμίσεων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα που μπορεί να γίνει Ταμείο Νομισματικό, όπω είπε ο Ρέμον από το πρόγραμμα του Ταμείου Εξυγείας των Τραπεζών και κάποιο Ταμείο Εγγύσεως των Καταθέσεων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλους ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη. Κατά λοιπά, οι δημοσιονομικές προτεραιότητες της ε, Ευρωζώνης διαφορετικές, η χρηματοδότηση ε, για την ε, μεταναστευτική κρίση, για την συνέπεια στις διασκέψεις των Παρισίων για το κλίμα, χρηματοδότηση της πολιτικής επενδύσεων του σχεδίου Juncker και δεν θα πρέπει να θυσιάσουμε τις προτεραιότητες αυτές προς όφελος ενός ονείρου που κάποια κράτη-μέλη μας βάζουν μπροστά στα μάτια για να μας κάνουν να δεχτούμε τη δημοσιονομική λιτότητα κατά τα λοιπά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Alfred Sand. Το πρόβλημα που έχω με το κείμενο ποιο είναι. Ξεπερνά τις πολιτικές έννοιες και τις ιστορικές τιάφτες στη συζήτηση. Οι τεχνοκρατικές προσεγγίσεις ίσως να είναι ενδιαφέρουσες, όμως χρειαζόμαστε πολιτική ανάλυση τώρα. Ποια είναι η κατεύθυνση της Ευρωζώνης, ποιος ωφελείται από τι και πού βρίσκονται τα δομικά προβλήματα. Η στατική είναι σαφέστατη μέσω μικρών τεχνοκρατικών βημάτων προχωράς και μετά σταδιακά φτάνεις στην κατάσταση που θα πρέπει να παγιωθεί. Πρέπει να υπάρχει πολιτικός ιδιασμός όμως. Θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα πολιτικών διαπραγματεύσεων των μελών της Ευρωζώνης, μεταξύ των μελών της Ευρωζώνης. Μιλάμε για φεντεραλισμό ουσιαστικά που δεν θέλει να ονομάζεται. Αυτό είναι λάθος λάθος να ακολουθούμε φεντεραλιστικό δρόμο χωρίς να ξεκάθαρο ότι χρειάζεται πλήρης πολιτική αποδοχή αυτού. Τεχνοκρατικές προσεγγίσεις δεν μπορούν να ομοιοποιηθούν μέσω των υφισταμένων δομών. Το Ευρωκοινοβούλιο, Φερρυπίν, δεν είναι ο θεσμός που μπορεί να ομοιοποιήσει ε, αυτό που κάνουμε δημοκρατικά. Και αυτό το βλέπουμε από τα αποτελέσματα των εκλογών και των δημοψηφισμάτων. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα που δεν εντοπίζεται, η πολιτική, οικονομική και διαφθορτική ανισορροπία που υπάρχει στην Ευρωζώνη μεταξύ κέντρου, Ανατολής Βοκενότου Και αν δεν αντιμετωπιστεί πολιτικός πώς και οικονομικός πώς, δεν θα βρούμε λύσεις που θα καταλάβει ο κόσμος. Ποιο είναι το θέμα. Θα έχουμε το πρόβλημα της σωστής επιστροφής των συνεισφορών. Γιατί να μην τεθεί επιτάπητος. Θα έπρεπε. Δομικά τώρα η Ευρωζώνη λειτουργεί σαν νομισματική ένωση που δεν λειτουργεί στο βέλτιστο βαθμό. Και θα μειώνεται η απόδοσή της ε, με την ε, παρουσίαση των προβλημάτων. Καλός ο σχεδιασμός, αλλά η πολιτική νομιμότητα και η πολιτική λογική για την Ευρωζώνη δεν ε, ευσταθούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νουβάκοφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι ειδικό, αλλά άκουσα, δεν είμαι γιατρός, αλλά άκουσα ότι το ευρώ είναι ασθένεια. Ε, είναι, κάτι, είναι ένα χάπι το ευρώ, πικρό, δύσκολο κατάπιωτο, αλλά είναι μια λύση. Άκουσα επικρίσεις ότι είναι λάθος ότι οι πλούσιες χώρες πρέπει να δίνουν πόρους στις στοχότερες της Ένωσης. Σωστό. Είναι η πολιτική συνοχής όμως αυτή. Βασικός πυλώνας της Ένωσης. Αν δεν συμφωνούμε από αυτού, θα πρέπει να θέσουμε τεράστιο θέμα για την ύπαρξη της ίδιας Ένωσης. Πιστεύω ότι κανένα μοναδικό νόμισμα συμπεριλαμβανομένης και της Ιταλικής Λιρέτας θα μπορούσε να ανταγωνιστεί άλλα ισχυρά νομίσματα στον κόσμο όπως το αμερικανικό δολάριο ή κάποιο άλλο νόμισμα. Το μέλλον λοιπόν ανήκει στο ευρώ. Έχουμε πολλά προς επίλυση προβλήματα. Το πρόβλημα που είχαμε στην Ελλάδα και έχουμε στην Ελλάδα είναι κίτρινη κάρτα που υψώνεται. Προειδοποίηση ότι πρέπει να λύσουμε όλα τα προβλήματα του νομίσματος. Ίσως η λύση είναι μια πλήρης τραπεζική ένωση, όχι όμως η δημιουργία κι άλλου άχθους οικονομικού ή φυσικού. Λοιπόν, πρέπει να δούμε ποια είναι τα προβλήματα του συστήματος, αλλά δεν πρέπει να σκοτώσουμε τον ασθενή, διότι έχει πυρετό, να του δώσουμε ένα χάπι του ασθενούς αυτή είναι η λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ντελάγκε. Η Άστη Ντελάγκε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολλά ήδη υπόθηκαν και βέβαια δεν είναι τέλεια η ΟΝΕ, άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να την ενισχύσουμε. Απλά ανησυχώ, γιατί έχουμε ένα πολύ κακό ιστορικό μέχρι τώρα. Αν δούμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το πάνε και πολλοί και όλες αυτές οι υποσχέσεις μεταρρυθμίσεων που έμειναν στα λόγια, οι στάσεις αναχώρα. Ανησυχώ λοιπόν ότι αν αρχίσουμε να οικοδομούμε κάτι καινούριο πάνω στις αποτυχίες του παρελθόντος ε, θα χτίζουμε παλάτια στην άμμο και τα κράτη-μέλη τελικά. Όταν εμείς μιλάμε για ενίσχυση της δεν θα πρέπει στα κράτη-μέλη να δείξουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι και να δείξουμε ότι μπορούμε να τηρούμε τις συμφωνίες μας και τις συνθήκες. Φυσικά τα κράτη-μέλη έχουν το μεγαλύτερο μερδίο ευθύνη, αλλά και εμείς από δικής μας πλευράς θα πρέπει να τα πούμε όλα αυτά ξεκάθαρα, ότι χρειάζονται υγιή και σταθερά θεμέλια, γιατί κατά το παρελθόν νομίζω ότι ε, αποδείχθηκε και παραδεχθήκαμε ότι αυτά τα θεμέλια έχουν ε, δομικές, ε, δομικά προβλήματα, δομικές αντιναμίες. Είπε κάποιος ότι πάνω απ' όλα χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση του ενωσιακού προϋπολογισμού. Αυτή είναι αφετηρία. Μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο πρέπει να αποδείξουμε ότι, για παράδειγμα, τα διορθωτικά μας ταμεία το Ταμείο Συνοχής που θα προετοίμασε τα κράτη-μέλη για να ε, προσχωρήσουν στην Ευρωζώνη. Θα μπορούσαν να προσφέρουν τόσο πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία να σχετίζονται πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα στις οικονομικές πολιτικές που είναι αναγκαίες για τις ε, χώρες μέλη της Ευρωζώνης, σε στάση αναχώρα. Ο Αλέλα Λαμασούρ ανησυχεί και το καταλαβαίνω ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο για οικονομικό θεματολόγιο ο προπολογισμό τη Ένωση, αλλά έχουμε και τη μετανάστευση, τη θέση τη Ευρώπη στον κόσμο, οικονομικό θεματολόγιο και βιωσιμότητα. Όταν μιλάμε για το οικονομικό σκέλο, να δούμε πρώτα πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ε, με μεγαλύτερη διασύνδεση στις διαθροτικές πολιτικές και με την πολιτική μας να ε, στηρίξουμε και να προασπίσουμε αυτές τις κόκκινες γραμμές στην οικονομική πολιτική. Αλλιώς όλα τα τόσο ε, μεγάλα όνειρα αν δεν ε, στηριχθούν πάνω σε γερά θεμέλια δεν θα είναι παρά ένας πυρός από τραπουλόχαρτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια έντονη συζήτηση. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να ακούσουμε σχόλια από τους εισηγητές αν θέλουν. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Και βεβαίως ε, το φάσμα των πολιτικών αξιολογήσεων νομίζω είναι παρόμοιο με αυτά τα οποία βρίσκει κανείς ε, σε μια ανάγνωση της ε, ανάλογης βιβλιογραφίας. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Εγώ άρχισα να ενδιαφέρομαι για την ευρωπαϊκή πολιτική στις σπουδέ μου τέλη 60-70 που τότε η ΕΟΚ είχε γνωρίσει μεγάλες αναταράξεις και με τι συνδέθηκαν όλα αυτά. Και τελικά κινδύνευε με διάλυση η ΕΟΚ και δεν ήταν τυχές οι εκθέσεις τότε και οι άλλες πρωτοβουλίες που στόχο είχαν να υπάρξουν κάποια σταθεροποιητικά στοιχεία. Όποιος θεωρεί λοιπόν τώρα πως ε, μπορεί να προβλέψει το τέλος του ευρώ γιατί θα γίνουν τα πράγματα καλά δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του απέναντι στους πολίτους. Και είμαστε σε ένα παγκόσμιο χωριό και είτε μιλάμε για τη Μάλτα είτε για τη Γερμανία, μόνος του δεν θα μπορέσει κανείς να σταθεί. Και εδώ πέρα συμφωνώ με τον Παουλ Τάγκ. Το θέμα του τίτλου είναι σημαντικό στο τέλος της διαδικασίας. Δεν πρόκειται για μέσα, πρόκειται για στόχους και δράσεις για ε, ένα διαρκή ε, μηχανισμό σταθεροποίησης της ε, Ευρωζώνης. Αυτό είναι το θέμα. Και η Εστέρ Ντελάγκη επίσης έχει δίκιο. Πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτά τα οποία έχουμε και τα λάθη του παρελθόντος. Και πρέπει να προσέξουμε πράγματι να μην χτίσουμε στην άμμο παλάτια. Και με βάση αυτή την ανάλυση πρέπει ταυτόχρονα να σκεφτούμε ποια είναι τα πρώτα που μπορούν να πάνε γρήγορα για να δοθούν κάποια μηνύματα, ότι μάθαμε δηλαδή κάτι ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι καινούριο χωρίς να παραμελούμε το ότι απαιτούνται νέα ενεργητικά βήματα. Αυτά νομίζω θα πρέπει να μπουν σε μια νέα μορφή με υπευθυνότητα. Και εδώ πέρα η κυρία Γκουλάρ έχει δίκιο. Πρέπει τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις να είναι στην πρώτη γραμμή αν είναι να είμαστε αξιόπιστοι. Και θα πάω παραπέρα από αυτό το οποίο είχα πει στην αρχή. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πράγματι υπέρ του ενιαίου προϋπολογισμού και δεν θα πρέπει συνεχώς να μετατοπίζονται εκτός του, Ευρωπαϊκού του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της εποπτείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διάφορα ταμεία και μηχανισμοί σταθερότητας. Από την άλλη όμως βλέπω πως όταν μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο και βλέπουμε πώς χρηματοδοτούνται αυτή τη στιγμή τα 440 δισεκατομμύρια και μιλάμε για δημοσιονομικές δυνατότητες οι οποίες θα πάνε σε συγκεκριμένους σκοπούς, δεν θα έχουμε έναν παράλληλο προϋπολογισμό, τότε ρεαλιστικά βλέπω πως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα χωρίς ε, να υπάρχει η ευθύνη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γιατί υπάρχουν αποφάσεις ε, του Συνταγματικού Δικαστηρίου που δεν μπορούμε να τις ε, παραμερίσουμε. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι συγκεκριμένο πρόβλημα μιας χώρας, αλλά δεν έχω καμία όρεξη να παραμελήσουμε αυτά τα πράγματα και μετά να ακυρωθεί το όλο το εγχείρημα. Γιατί το θέμα είναι και το θέμα του κοινοβουλευτισμού και στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί πού ε, βρίσκονται τα εθνικά κοινοβούλια σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν περιορισμένο ρόλο και είμαι ευγενικός. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρόλα του τα ελλείμματα είναι το μοναδικό άμεσα ερετό θεσμικό όργανο Οπότε θα πρέπει να οδηγηθούμε πράγματι σε ένα μηχανισμό σταθερότητα, όχι όμω σε έναν ανταγωνισμό με τα εθνικά κοινοβούλια. Πρέπει να υπάρξει ένα επαγγελματισμό τη συνεργασία μα. Τώρα δεν θέλω να φτιάξουμε καινούρια θεσμικά όργανα. Υπάρχουν κάποιε λύσει ενδιάμεσε, αλλά χωρί να αναλάβει την ευθύνη του και το εθνικό επίπεδο όσον αφορά τους πόρους, το θέμα της συναπόφασης, δεν θα επιτύχουμε τους ε, στόχους μας και πρέπει να το πούμε αυτό ειλικρινά. Η κυρία Χιούμπνερ είπε πως πρέπει να δώσουν περισσότερα κίνητρα αντί για αντικίνητρα. Ναι, εγώ είμαι υπέρ των κινήτρων. Α, είμαι υπέρ και της ατομικής ευθύνης. Μόνο έτσι υπάρχει μετά απέτηση για αλληλεγγύη. Αυτό δεν αποκλείει όμως ότι κάποια στιγμή υπάρχουν υποχρεώσεις και πιθανώς και κυρώσεις. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Δεν είναι μόνο θέμα χωρών. Αυτό αφορά και τις σχέσεις ε, πόλεων και εθνικών κρατηδίων ε, εντός μιας χώρας κτλ. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην εξισορρόψη αυτών των δύο. Αλλιώς δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Και βεβαίως ξεκάθαρο ότι οι πυλώνες στην έκθεση ήδη ε, πρέπει να έχουν ε, την ίδια αξιολόγηση όπως αναφέρει και η έκθεση των πέντε πρόεδρων. Και η Κομισιόν κάποια στιγμή πρέπει να δώσει βάση. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε στο πέμπτο βήμα πριν από το δεύτερο και να ενοχλούνται τα κράτη-μέλη. και να σέρνουν τα πόδια τους και να μην εφαρμόζουν τα συμφωνημένα. Γιατί βεβαίως, αυτό μας δυσκολεύει μετά όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Ευχαριστώ, euh, euh, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω να πηχήσω τα υποθέντα. Αυτό το πετύχω μέσω πέντε βασικών προβληματισμών. Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το βασικό μήνυμα του, του, της εκθέσεως. Ο πρόεδρος κ. Σαχτουή είπε ότι πρέπει να απευθυνθούμε στους Ευρωπαίους. Βεβαίω. Όμως πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να στέλνουμε ένα μήνυμα σαφές προς το Συμβούλιο. Διότι γνωρίζουμε ότι όλες οι πρωτοβουλίες αναφέρθηκαν σε πανεπιστημιακές γνώσεις και θέλουμε να δούμε αν χρειαζόμαστε προπολογισμό τη Ευρωζώνης. Παρόλο που Αλέων Λαμασούρα αμφισβήτησε αυτή την ιδιαιτερότητα αυτού του προπολογισμού τη Ευρωζώνης. Έχουμε τους 4 τους 5 προέδρους, προτάσεις, αντιπροτάσεις κλπ. Και όλα λένε ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να στείλει μήνυμα στον αφορά αυτό. Όχι μόνο στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, αλλά και στους υπουργούς οικονομικών. Τι θέτε το εξή λοιπόν. Δημιουργείται ηθικός κίνδυνος. Πώς μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Και έρχομαι στο δεύτερο στοιχείο που θέλω να αναφέρω. Δεν αγνώ ότι κάποιες πτυχές των προτινομένων απαιτούν τροποποίηση των συνθήκων. Ε, μπαίνουμε όμως έτσι σε μια άλλη έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι έργο που μοιράζονται έκθεση Μπορκ Μπορ-πρεσό και έκθεση Βερχόφστατ. Για μας τίθεται ένα ερώτημα λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Τι χρειαζόμαστε, ούτως ώστε να λειτουργούν όλα τον καλύτερο τρόπο να μην έχουμε μεγαλύτερη ενεργεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποκλήσεις ε, μεταξύ των χωρών. Για να το καταφέρουμε αυτό. Όπως προτείνει ο Αλφέτ Σαντ, να ασκήσουμε κάποιο φεντεραλισμό και να φύγουμε από τη μέθοδο των μικρών βημάτων. Και ο Μπάς Εκχάουτ ανησυχούσε γι' αυτό. Για τα συνεχή μας τορέματα που απαιτούνται για να δημιουργηθούν τα αναγκαία μέσα. Έτσι που τίθεται το θέμα, οδηγούμεθα προς κάποιες διευκρινήσεις. Και τελικά προσπαθούμε να βρούμε τι λείπει από την Νομισματική και Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, που είναι ο προπολογισμό της Ευρωζώνης, όσον αφορά τον ηθικό κίνδυνο. Κάτι που αναφέρθηκε. Απηχώ αυτά που ακούσαμε και στην ακρόασή μας. Το θέμα του ηθικού κινδύνου είναι σημαντικό, πρέπει να ληφθεί ε, υπόψη, αλλά δεν θα πρέπει να αποτελέσει επιχείρημα για δράνεια. Καμιά φορά θεωρούμε ότι το παίζουμε σαν χαρτί, σαν τζόκερ, για να θέτουμε βέτο σε κάθε πρόταση και δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Τρίτο στοιχείο. Για να κάνουμε τι με τον προβλησμό της Ευρωζώνης, υπάρχει ένα δημόσιο αγαθό της Ευρωζώνης. Το έθεσε ο Αλένα Μασούρ και άλλοι, παρατηρώντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η Ευρωζώνη. Τι βλέπουμε. Έχουμε ιδιαιτερότητε οικονομικές. Το παρατηρήσαμε αυτό. Μειώνεται το βάρος του αυτόματου σταθεροποιητού, αυξάνεται η απόκληση μεταξύ των οικονομιών και έχουμε πολύ χαμηλό επίπεδο επενδύσεων κάτω από το επίπεδο επενδύσεων τη υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και αυτά είναι ιδιαιτερότητε τη Ευρωζώνη που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να συζητήσουμε τι δυσκολίε για να εμβαθύνουμε. Αυτό το ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, πώ θα μετατρέπεται σε συγκεκριμένε επενδύσει. Οι διασυνδέσει ιδεοδρομικέ περίπου μεταξύ Λισαβόνα, Βερολίνου ή Παρισίων και Βερολίνου είναι ένα, ε, κάτι που αφορά την Ευρωζώνη, ένα κοινό αγαθό τη Ευρωζώνης, δεν νομίζω. Υπάρχει διάκριση μεταξύ λειτουργία και κανόνων λειτουργία της Ευρωζώνης και τι παράγει μακροοικονομικό για την Ευρωζώνη και απ' την άλλη συγκεκριμένα κοινά αγαθά όσον αφορά τις επενδύσεις. Τελευταίο σημείο. Προπολογισμό Η θέση του Ευρωκοινοβουλίου πάντα ήταν ότι ο Ευρωπαϊκό μηχανισμός σταθερότητας ε, πρέπει να οδηγεί ε, στη σταθερότητα. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μηχανισμό όμως που θα παγιδεύεται από τους κανόνες του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Διαφορετικά, αν το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ασύμετρους κλειδονισμούς. Είναι μια λεπτομέρεια που θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά. Τέλος, Συμφωνώ απόλυτα με τον Ράιμερ Μπέργκερ για τα εθνικά κοινοβούλια και τη συμμετοχή τους. Πρέπει να επαγρυπνούμε από αυτού και να είμαστε πολύ απαιτητικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημαντικότητα τη συζήτηση. Σημειώθηκε κάποια πρόοδος. Διαπιστώθηκαν και διαφορές. Αλλά και στοιχεία συγκλήσεως Πρέπει να συζητήσουμε τους στόχους και τη λειτουργία πέρα από τα μέσα. Εντοπίζουμε ειδικέ λειτουργίες που συνδέονται, ιδιαίτερε λειτουργίες που συνδέονται με το κοινό νόμισμα, ιδιαιτερότητες. Να μην υπάρχει επικάλυψη με τις ευρύτερες λειτουργίες της Ένωσης. Μιλάμε για ένα εργαλείο για την Ευρωζώνη, αλλά όπως και η Τραπεζική Ένωση μπορεί να είναι ανοιχτό σε συμμετοχή απο κάτι κράτη-μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Υπάρχει και η δυνατότητα ειδικού εργαλείου που θα πρέπει να εδράζεται επί του προϋπολογισμού, του σχετικού πλαισίου του προϋπολογισμού και του ευρώ. Μπορούμε να έχουμε πολυεπίπεδη ένωση, πιστεύω, εντός του κοινού νομικού πλαισίου. Αυτό είναι σημαντικό σαν στοιχείο. Μετά και κάτι άλλο. Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες του ηθικού κινδύνου, κυρώσεων και κινήτρων, πρέπει να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση της νομισματικής ενώσεως. Διεφάνισαν λοιπόν αρχές, επί των οποίων επετέθη κάποια σύγκληση. Άρα, μπορούμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες των ζητημάτων που έθεσαν οι εισηγητές. Ζω, θες να πεις κάτι? Χαίρομαι γιατί η συζήτηση αυτή ήταν πολύ πλούσια και διασκεδάστηκαν κάποιε παρανοήσει, Φυσικά και δεν φέρνουμε αντιμέτωπε στις χώρε τη Ευρωζώνη με τι χώρε τη υπόλοιπη τη Ένωση. Αλλά αυτό που είναι σαφέ είναι ότι όταν υπάρχει δυσκολία σε κάποια από τις χώρες της Ευρωζώνης και χρειάζεται το χρέος, το περιβολικό κάποιας χώρας ε, να καλυφθεί ε, συλλογικά. Δεν θα πρέπει να συμμετέχουν 28 χώρες μέλη μέσω του μηχανισμού σταθερότητας, αλλά οι χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Και βέβαια τα εθνικά κοινοβούλια είναι σημαντικό να συμμετάσχουν γιατί θα πρέπει άλλωστε και να ψηφίσουν τις απαραίτητε πιστώσεις. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ίσως είναι κατά την άποψή μου ε, ένας προθάλαμος, ε, μία πρώτη εκδοχή εφόσον ουσιαστικά ε, το χρέος των ε, χωρών της Ευρωζώνης. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι το πρώτο βήμα πριν από ένα προπολογισμό της Ευρωζώνης. Για τον τίτλο τώρα που είπατε, Δύσκολο ήταν και να βρεθεί ένα τίτλο, αλλά καλό είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι εργασίε και μετά θα βρούμε ίσω και τον πιο κατάλληλο τίτλο. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίαση των Επιτροπών ΕΚΟΝ και ΜΠΑΤΣ και προχωρούμε στη συνεδρίαση, την τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Ε, διάλειμμα ένα λεπτό για να αποχωρήσουν όσοι δεν πρέπει να παραμείνουν.